Okay, good morning. Let's start. Ε, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε. Σας καλωσορίζω στη συνεδρία της Επιτροπής Αναφορών. Ισπανιόλ. Θα μιλήσω ισπανικά. Καθώς υπάρχει διερμηνία. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο σημείο. Uh, del έγκριση το σχεδίου της ημερησίας διάταξης. Ε, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, μπορεί να εγκριθεί το σχεδίο ημερησίας διάταξης. Ε, επομένως, εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται. Περνάμε στο σημείο 3, έγκριση των πρακτικών τη συνεδρίαση 4η και 5η Σεπτεμβρίου 2019. Τα πρακτικά έχουν μοιραστεί σε όλα τα μέλη τη Επιτροπή. Και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, που από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν, θεωρούμε ότι εγκρίνονται ανακοινώσεις της Προέδρου δεν υπάρχουν. Περνάμε στο σημείο 5 που είναι έκθεση σε σχέση με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Διευθυνσολαβήτριας κατά το 2018. Ο κύριος Γιάρ είναι ο εισηγητής και έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Δημοσιολογητή. Θέλω να σας πω το εξή οι πολίτες μπορούν βεβαίως σε περίπτωση παραβίασης των ε, δικαιωμάτων, του τους να απευθύνονται στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια και ακριβώς επειδή και η Επιτροπή Αναφορών έχει παρόμοια δραστηριότητα, είναι προφανές ότι έχουμε πολύ στενή σχέση. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία, Ράιλ, την κυρία Οράιλη για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε το 2018. Όπως γνωρίζουμε, το Δεκέμβριο στην Ολομέλεια δεν θα ψηφιστεί μόνο η ετήσια έκθεση της ε, διαμεσολαβήτριας, αλλά θα ε, ψηφιστεί και ο νέος Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ή η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια. Γι' αυτό και προσπάθησα να συντάξω ένα ισορροπημένο κείμενο και ελπίζω να τύχει και της υποστήριξη των συναδέλφων, ώστε η Επιτροπή Αναφορών να μην ε, γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης παράπλευρων πολιτικών διαμαχών. Εγώ θεωρώ ότι η Ευρωπαία διαμεσολαβήτρια γίνεται όλο και πιο ορατή στους Ευρωπαίους πολίτες. 490 έρευνες έκανε η διαμεσολαβήτρια το 2010, ε, διαμεσολαβήτρια, διαφάνεια, πρόσβαση σε δημοσία έγγραφα, ήταν τα αντικείμενα που την απασχόλησαν. Ε, ιδίως αξιοσημείωτη είναι η δουλειά που έκανε η διαμεσολαβήτρια στο ζήτημα της έλλειψης διαφάνειας στο Συμβούλιο, ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει και εδώ στην Επιτροπή μας. Ε, πολλές φορές η αποφάση του Συμβουλίου είναι ένα μαύρο κουτί που δεν γνωρίζουμε κι εμείς ακόμη ως Ευρωβουλευτές για ποιο λόγο και με ποιον τρόπο έχουν ψηφίσει συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Η διαμεσολαβήτρια θεωρεί ότι αυτό πρέπει να αλλάξει συμφωνούμε και εμείς και θεωρούμε ότι πραγματικά ε, και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αυτό το ζήτημα της έλλειψης διαφάνειας στο Συμβούλιο. Χαίρομαι λοιπόν για τη συνεργασία που είχαμε με τους συναδέλφους ε, για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης. Σημαντικές ημερομηνίε που επίκυνται είναι για τις τροπολογίες 7 Οκτωβρίου, δηλαδή σχετικά σύντομα, από 21 Οκτωβρίου ε, εκείνη την εβδομάδα κάποια στιγμή θα γίνει η συνεδρία Σκιωδών, διότι θα γίνει και τον Δεκέμβριο η ψηφοφορία στην Επιτροπή Πέτη και αν με έχουν ενημερώσει σωστά μπορεί ε, απευθείας η έκθεση να πάει και στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Ξαναλέω, χαίρομαι πάρα πολύ για τη συνεργασία που είχαμε μέχρι στιγμή, για την συνεργασία που επίκειται να έχουμε τι επόμενε εβδομάδε και ε, ε, πάμε και στην ψηφοφορία. Ε, ευχαριστώ κύριε Γιάρ. 7 Οκτωβρίου στις 3 το απόγευμα λίγη η προθεσμία υποβολής ε, ετοιμάτων τροπολογιών. Κύριε Εύη. Ευχαριστώ. Θέλω να σχολιάσω το σχέδιο κειμένου του κυρίου Γιάρ. Τον ευχαριστώ, όμως ε, ήθελα να τονίσω κάποια σημεία με τα οποία δεν συμφωνώ. Διαφωνώ κυρίως ε, στην αναφορά που γίνεται για την απόφαση του δικαστηρίου του 2018 γιατί αναφέρει ο συνάδελφος ε, τα συμπερίσματά της επίσημα, αλλά δεν ε, αναφέρει ε, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι προέκυψε σχετικά με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την απόφαση. Αναφέρεται ότι οι αρχές της διαφάνειας ε, και της δημοσιοποίησης είναι εγγενείς στην ε, νομοθετική διαδικασία της Ένωσης. Δηλαδή θα πρέπει οι πολίτες να μπορούν να παρακολουθούν τη διαδικασία, να μπορούν να συμμετέχουν και να έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες. Και εγώ νομίζω ότι είναι καλό να το υπογραμμίζουμε αυτό, γιατί σε άλλα σημεία του κειμένου και συγκεκριμένα σε σχέση με το ρόλο και τις δραστηριότητες ε, που έχει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ και του ε, Προέδρου της ε, γίνεται αναφορά στην ελευθερία τους να αποφασίσουν αν θα συμμετέχουν σε διάφορες συζητήσεις ακόμη και κλεισμένων το θυρών. Αυτό αν εγγυάται την καλύτερη διεξαγωγή της νομισματικής πολιτικής. Όμως αυτό έρχεται σε μεγάλη αντίθεση ε, με τις νομικές αναφορές στην απόφαση αλλά και τις ίδιες τις συστάσεις της διαμεσολαβήτριας. Γιατί στην περιπτωση Draghi Ντράγκη G30 είχε υπογραμμίσει η διαμεσολαβήτρια ότι μη διαφανείς συμπεριφορές ε, πρέπει να καταδικαστούν. Και ε, κάτι ακόμη για τις ε, συνεδριάσεις ε, όπου συμμετέχουν ή οργανώνονται από τράπεζες υπό την εποπτεία της ΕΚΤ. Και δύο άλλα πράγματα, πολύ γρήγορα. Διαφωνώ στα σημεία που αναφέρονται στις δραστηριότητες άσκησης πίεσης, lobbying. Γιατί και πάλι αναφέρεται σε διοργανική συμφωνία ο συνάδελφος, ενώ εδώ στο Κοινοβούλιο Έχουμε ζητήσει πολλάκις να φτάσουμε σε ένα νομοθέτημα που να είναι νομικά δεσμευτικό και υποχρεωτικό. Όχι μόνο για τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για όλα τα τρίτα μέρη. Ε, νομίζω ότι ήρθε λοιπόν η στιγμή να ζητήσουμε για νοιαστή φορά, με δυνατή φωνή, να αναθεωρηθεί ο οργανισμός του 2001-1049, ε, ο οποίος θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Κύριε Άουκεν. Ευχαριστώ, Πίτερ. Πολύ καλή έκθεση αυτή. Χαίρομαι που αναγνωρίζεις το έργο της κυρίας Οράιλη. Και αναφέρεις ότι έχει βελτιώσει την ε, παρουσία, τη δημόσια παρουσία ε, του διαμεσολαβητή και ότι αποτελεί πραγματικά εγγύηση ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υιοθετήσαμε το καινούριο καθεστώς που διέπει τη λειτουργία του διαμεσολαβητή και κρεμίζει ενώπιον του Συμβουλίου το κείμενο αυτό. Ε, κάποιοι δεν το κατάλαβαν πολύ καλά. Εμείς έχουμε την ευθύνη για το διαμεσολαβητή. Δηλαδή, εμείς κάναμε τη δουλειά μας, αλλά αυτό δεν αποτελεί απλώς ένα ψήφισμα. Αυτή η δουλειά δεν είναι ένα απλό ψήφισμα. Ο κανονισμός που διέπει το διαμεσολαβητή είναι δική μα αρμοδιότητα. Εμείς ψηφίσαμε τον κανονισμό. Αυτά που λέει ο προηγούμενος πρόεδρος δεν έχουν καμία σχέση με τη θέση του Κοινοβουλίου. Δεν πρόκειται για ένα απλό ψήφισμα. Ήταν ε, μεγάλο σοκ για μένα αυτό. Αλλά τέλος πάντων το λέω εν παρόδο. Θα πρέπει να πιέσουμε για το θέμα της διαφάνειας στο Συμβούλιο. Η κυρία Τόμ και ο κύριος Λάινεν ε, απάντησαν πολύ σαφώς στην έκθεση του ε, διαμεσολαβητή. Δεν είναι δύσκολη η έκθεση, να διαβαστεί η έκθεση της διαμεσολαβήτριας, είναι μόνο 13 σελίδες. Κάποιοι φοβούνται να τη διαβάσουν, αλλά αυτό που σημαίνει στο Συμβουλίο παραβαίνει τη συνθήκη. Η συνθήκη δίνει το δικαίωμα στους πολίτες να παρακολουθούν την νομοθετική διαδικασία. Αν δεν μπορούν να παρακολουθήσουν την κυβέρνησή τους, ε, ε, παραβαίνουμε τη συνθήκη. Δεν μπορεί οι πολίτες να γνωρίζουν μόνο για το αποτέλεσμα της διαδικασίας. Χαίρομαι που στηρίζεται η άποψη της κυρίας Οράιλη να επιμείνει Αν ξεκινήσει ο τριμερής διάλογος χωρίς να ανοίξουν διαδικασίες του Συμβουλίου, τότε διευκολύνουμε το ρόλο των λομπιστών να πιέζουν το Συμβούλιο. Και συμφωνώ και για αυτά που είπατε για την τράπεζα. Ευχαριστώ, Πίτερ. είναι σημαντικό εμείς, ε, η δική μας Επιτροπή, να κρατήσει ψηλά τον πύχη. Thank you, Mr. Um, Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τέρες. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει στην έκθεση αυτή. Ως ε, σκιώδης των σοσιαλιστών μπορώ να σας πω από τώρα ότι θα υποβάλουμε κάποιες τροπολογίες. Απλά σου θέλω να επισημάνω κάποια ζητήματα. Πρώτον, ε, χαιρετίζουμε και εκτιμούμε την δραστηριότητα της ε, διαμεσολαβήτριας ε, για το ζήτημα της διαφάνειας, λογοδοσίας και της προτιμώσας πρόσβασης σε έγγραφα καθώς και της ε, διαδικασίας fast track που ξεκίνησε. Θεωρώ ότι οι δραστηριότητες της έχουν διευκολύνει τους Ευρωπαίους πολίτες και τη σχέση τους με, ε, με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτό βοήθησε στην ε, βελτίωση τη εικόνας των ε, θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μάτια των πολιτών. Εμείς εγκρίνουμε και τις συστάσεις και χαιρετίζουμε τις συστάσεις της διαμεσολαβήτριας προς το Συμβούλιο. Θεωρούμε και εμείς ότι το ζήτημα της διαφάνειας είναι σημαντικό όχι μόνο στο Συμβούλιο αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι η εστίαση της έκθεσης ε, στο ζήτημα του, των λόμπι πρέπει να ενισχυθεί. Αλλά, όπως είπα, θα υποβάλουμε και κάποιες σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ, κύριε Τόμ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ε... Αν είσαι έκτος, δεν σου μένουν και πολλά πράγματα να πεις. Τα έχουν πει προηγούμενοι. Καταρχάς να ευχαριστήσω και εγώ τον Πέτερ για την εξαιρετική προσπάθεια του. Δεν συμβαίνει και πολύ συχνά να τον υποστηρίζω πλήρω. Ε, να που συνέβη και αυτό. Εγώ δύο τροπολογίες σκέφτομαι να υποβάλω. Θέλω να αναφερθώ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που ε, ε, ε έλαβε σύσταση από την ε, κυρία Οράιλη να, να χειριστεί καλύτερα το ζήτημα της ισότητας των φύλων και ε, και για το ζήτημα των, ε, της διαφάνειας των θεσμικών οργάνων θεωρώ ότι σωστά το έχει θέσει το θέμα για την ε, περίοδο ε, cooling down την τριετή. Εμείς θέλουμε να ε, ξεκαθαρίσουμε ότι όταν λαμβάνεται μια απόφαση δεν είναι δυνατόν αυτή να ξεχνιέται μετά από έξι μήνες. Βεβαίως αυτά τα ζητήματα ε, δεν, μπορούμε να τα χειριστούμε όλα μέσω μιας έκθεσης, αλλά παρόλα αυτά καλό είναι να αναφέρονται και εδώ. Ευχαριστώ Πέτερ σε κάθε περίπτωση για την καλή συνεργασία που είχαμε. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, Θέλω και εγώ καταρχάς να ευχαριστήσω τον ε, συνάδελφο Γιάρ. Πρόκειται για μια έκθεση η οποία ε, δεν είναι εύκολο να τη συντάξει κανείς. Θα υποβάλουμε και εμείς ε, κάποιες τροπολογίες. Είχαμε κάνει και μια σχετική συζήτηση με τον κύριο Γιάρ. Και πράγματι είχαμε συμφωνήσει ότι είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της διαφάνειας στο Συμβούλιο. Όμως θα πρέπει να δούμε λίγο και τα δικά μας τα του οίκου μας. Γιατί υπάρχουν λόμπι τα οποία δραστηριοποιούνται και εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε και εδώ θα πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια. Στην τελευταία κοινοβουλευτική θητεία, για παράδειγμα, είχαμε έναν προβληματικό ε, ευρωβουλευτή στην Επιτροπή Γιούρι. Η υπόθεση κατέληξε σχεδόν στα δικαστήρια. Ε, η Γιούρη επίσης ε, αυτή τη στιγμή ε, έχει ελέγξει ζητήματα που σχετίζονται με την καταλληλότητα των οριστέντων επιτρόπων. Εκεί έχουν ακουστεί ζητήματα όμως τα οποία είναι πάρα πολύ ανησυχητικά αλλά ζητήματα που σχετίζονταν με την σχέση των οριστέντων επιτρόπων με ε, λόμπι, εκεί δεν ακούστηκαν επαρκή επιχειρήματα και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν κάποιοι υποψήφοι ε, να διαπιστωθεί ότι είχαν ε, κάποια σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά ε, παλαιότερες θέσεις που κατήχαν. Χωρίς όμως αιτιολόγηση, χωρίς καθόλου αποδεικτικά στοιχεία έγινε όλη αυτή η διαδικασία. Επρόκειται για μια τελείως αδιαφανή διαδικασία. Και αν ε, υποβάλω τροπολογίες για την έκθεση του κυρίου Γιάρ, ε, ακριβώς αυτό θα είναι το θέμα. Η Επιτροπή. Παρακαλώ, εκπρόσωπος Επιτροπής έχει το λόγο. Καλημέρα σας. δεν θα σχολιάσουμε στο στάδιο αυτό. Φυσικά θα περιμένουμε τις τροπολογίες και το τι θα ακολουθήσει για να πούμε πόσο καλά αξιολογούμε τη δουλειά σας. Σας ευχαριστώ. Πίτερ, θες το λόγο για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Ε, απλώς να ευχαριστήσω και εγώ τους συναδέλφους που έχουν συμμετάσχει στη συζήτηση αυτή. Ε, θα διαπιστώσατε κι εσείς ότι δεν υπάρχουν μόνο προθεσμίες ε, για τις τροπολογίες, υπάρχουν και άλλες ε, ημερομηνίε που επίκυνται. Σας ευχαριστώ φυσικά για την πρόθεσή σας να υποβάλλετε τροπολογίες. Έχουμε όμως ορίσει και συνεδρίαση των σκιωδών συντονιστών. Ε, νομίζω ότι πρέπει εν ώψη και της εκλογής της νέας δημοσιολογητρίας ή του νέου δημοσιολογητή να καταφέρουμε να καταρτήσουμε μια καλή έκθεση. Χαίρομαι για τη συνεργασία που θα έχουμε. Νομίζω ότι η έκθεση θα είναι καλή. Στο τέλος να γίνει η ψηφοφορία το Νοέμβριο εδώ στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια τον Δεκέμβριο και να τελειώσει το θέμα. Ευχαριστώ πολύ, Πίτερ. Να υπενθυμίσω ότι στι 7 Δεκάτου, στι 3 το μεσημέρι, έχουμε την προθεσμία κατάθεση τροπολογιών και ψηφοφορία στην Επιτροπή μα θα γίνει στι 12 Νοεμβρίου. Να περάσουμε στο έκτο σημείο της ημερική διάταξης. Έχουμε διάφορες αναφορές. Την 672, 673, 674... Όλες ε, είναι αναφορές που έχουν παρουσιαστεί από Ρουμάνους πολίτες σε σχέση με την ατμοσφαιρική ρήπανση στο Βουκουρέστι σχετικά με την ατμοσφαιρική ρήπανση στο χωριό υγειονομικής ταφής Ρουντένη στο Βουκουρέστι. Οι αναφέροντες δεν είναι παρόντες, αν δεν κάνω λάθος. Και επομένως, θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Αλεξάνδρα Ιμαντόμπρα. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ η Επιτροπή θα ήθελε να γνωστοποιήσει στο Κοινοβούλιο ότι υπάρχουν πολλές διαδικασίες σε ό,τι αφορά την διαχείριση των αποβλήτων στη Ρουμανία. Καταρχήν έλαβε δράση σε ό,τι αφορά το κλείσιμο 68 χωματερών λήφθη μία απόφαση πέρσι στην 1η Οκτωβρίου η Κομισιόν από τη Δικαιοσύνη και σήμερα η Κομισιόν εκτελεί την απόφαση αυτή. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνά και το να κλείσουν 101, 101 χώροι υγειονομικής ταφής ε, του Δήμου έπρεπε να κλείσουν μέχρι τις 16 Ιουλίου 2017 αυτή η χώρη υγειονομικής ταφής για αυτούς τους δύο φακέλους η Επιτροπή προβαίνει στην εκτέλεση των αποφάσεων και ε, αν δεν κλείσουν αυτοί οι χώροι, υγειονομική ταφή, ή δεν ε, ε, δούμε να κλείσουν αυτοί, αυτές οι 101 χωματερές, η Κομισιόν θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Σε ό,τι αφορά τώρα τη ρήπανση στο Βουκουρέστι το 2016, ξεκίνησε ένας πιλωτικός φάκελος. Τώρα, ερευνούμε σε ποιο βαθμό αυτές ε, οι χωματερές στο Ροντένι και στην Κιάζα πράγματι ρηπαίνουν την ατμόσφαιρα. Λήφθησαν ε, πολλά μέτρα ε, από την Επιτροπή σε σχέση με αυτούς τους χώρους υγειονομικής ταφής σε ό,τι αφορά τον διαχειριστή, την Ήριντεξ, Ένα μέρος των κελιών έχουν κλείσει, το C1 και το C5 και η δραστηριότητα λοιπόν ε, μειώθηκε γιατί έχουμε λειτουργία με δύο κελιά λιγότερα. Το 2016 επίσης μία άλλη περιβαλλοντική αρχή ε, συγγνώμη, μια άλλη άδεια δόθηκε ε, σε αυτόν τον διαχειριστή. Τώρα, έχουμε ουσιαστικά μία υπόθεση που εκκρεμεί στο δικαστήριο για την ακύρωση αυτής της άδειας. Η Κομισιόν παρακολουθεί αυτή τη διαδικασία ε, βάσει των πληροφοριών που έχουμε από την πύλη δικαιοσύνης της Ρουμανίας. Ε, έχουμε ε, τη ε, διαδικασία αυτή να βρίσκεται στο στάδιο της διοικητικής εξέτασης. Από τις πληροφορίες που έχουμε η εμπειρογνωμοσύνη θέλει να θεσπίσει σε ποιο βαθμό η περιβαλλοντική άδεια θα πρέπει να περιλαμβάνει και σε τιμές για το υδρόθιο αλλά και για άλλες ουσίες γιατί το υδρόθιο δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε ό,τι αφορά την ποιότητα του αέρα. Και ε, στο βαθμό που τα εθνικά δικαστήρια αποφασίσουν ότι πράγματι αυτή η άδεια δεν έπρεπε να έχει δοθεί, τότε οι ρουμανικές αρχές θα πρέπει να εκτελέσουν την απόφαση. Επίσης, στις συνεδριάσεις που είχαμε τον Ιούλιο του 2019 με την εισαγγελία μας ενημέρωσαν οι ρουμανικές αρχές ότι τα τελευταία ε, κοιλιά το πρέπει να κλείσουν μέχρι το 2020. Ε, η Κομισιόν λοιπόν είπε στη Ρουμανική κυβέρνηση μέχρι το τέλος αυτού του έτους να παρουσιάσει μια εναλλακτική λύση σε σχέση με αυτούς τους χώρους υγειονομικής ταφής ε, στα βόρεια του Βουκρεστίου. Και βάσει της ανακοίνωσης της Επιτροπής του 2016, ενώ εκρεμεί η υπόθεση στα εθνικά δικαστήρια, αυτά είναι σε καλύτερη θέση να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την επιδιόρθωση της κατάστασης. Επομένως, εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το πώς ανταποκρίνονται οι ρουμανικές αρχές. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Οι πολιτικές ομάδες θέλουν το λόγο. Δεν νομίζω ότι είχε ζητήσει κανεί το λόγο. Ο κύριος ε, Είμαστε, είμαστε, στο σημείο 6, έτσι. Προτείνω όλα αυτά, τα, όλες αυτές οι αναφορές να μείνουν ανοιχτές. Γιατί είναι σημαντικές οι ανησυχίες των ετούντων, των αναφερόντων. Το 7, θα περάσουμε στο 7 τώρα. Ωραία, θα κρατάω τα σχόλιά μου για αργότερα. Πρόεδρος. Α, κυρία Τόμ, δεν έχει πάρει το λόγο. Ε, συμφωνώ με την προηγούμενη πρόταση. Θέλω όμως να ρωτήσω την Κομισιόν το εξής. Είπατε ότι τα θέματα αυτά εκκρεμούν στα εθνικά δικαστήρια. Ξέρετε περίπου πόσο θα πάρει. Μιλάμε για χρόνια ή για μήνες μπροστά μας. Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας αυτών των διαδικασιών. Κοιτάξτε, ξεκίνησε το 2018 η δικαστική διαδικασία όταν ε, δόθηκε αυτή η περιληπτική άδεια, όμως ε, έχει ε, αν ζητηθεί και μια έκθεση εμπειρογνωμοσύνης μπορεί και να διαρκέσει. Δηλαδή αυτό δεν εξαρτάται από τις εθνικές δικαστικές αρχές, αλλά από τους εμπειρογνώμονες να συντάξουν την ε, έκθεση αυτή. Θα εκτιμούσαμε ότι θα μπορούσε η διαδικασία να τελειώσει και του χρόνου, αν ε, δοθεί αυτή η έκθεση εμπειρογνωμοσύνης. Γιατί ξέρετε, τώρα μια τέτοια έκθεση εμπειρογνωμοσύνης είναι ιδιαίτερα σκόπιμη σε τέτοιες υποθέσεις. Πρόεδρος, ευχαριστώ ακούσαμε την Κομισιόν και τα μέλη της Επιτροπής, οπότε θα κρατήσουμε ανοιχτές αυτές τις αναφορές. Παρακαλούμε να συνεχίσει η Κομισιόν την παρακολούθηση της κατάστασης και να μας ενημερώσει για τα όσα θα λάβουν χώρα ε, τώρα μετά από ένα χρόνο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που μας είπε η Κομισιόν. Περνάμε στο σημείο 7, 0581, ε, από Ρουμάνο Επίκο για τις ε, υποτιθέμενες παρατυπίες σχετικά με τη συλλογή και την καύση επικίνδυνων ιατρικών ε, αποβλήτων στη Ρουμανία. Δεν είναι εδώ αναφέρον, οπότε δίνω το λόγο ξανά στην Κομισιόν. Εδώ μιλάμε περίπου για το ίδιο πρόβλημα σε αυτή την, το υγειονομική υγειονομικής ο αναφέρον ε, καταγγείλει ότι είχαμε και ιατρικά απόβλητα. Η Κομισιόν απευθύνθηκε στι Ρουμανικέ Αρχές. Από ό,τι φαίνεται δεν αποτίθεται ιατρικά απόβλητα εκεί. Επίσης, μέσω τη ε, περιβαλλοντική ε, άδεια του 2019 η εταιρεία δεν δικαιούται να εναποθέτει τέτοια απόβλητα. Δεν έχουμε άλλε πληροφορίες σε σχέση με αυτό το θέμα. Δεν ε, υπάρχουν ε, εκεί λοιπόν ε, ιατρικά απόβλητα που εναποτίθεται σε αυτή την χωματερή, σε αυτό το χωρίο υγειονομική ταφή. Μιλάμε μόνο για απόβλητα που δεν είναι επικίνδυνα. Θα πρότεινα λοιπόν στο Κοινοβουλίο να χειριστεί από κοινού αυτή την αναφορά μαζί με τις αναφορές του σημείου 6. Uh, uh, και εγώ πιστεύω ότι αυτά τα δύο θέματα θα πρέπει να ενοποιηθούν γιατί μιλάμε ουσιαστικά για την ίδια εταιρεία που ρηπαίνει και παρακαλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το θέμα προσεκτικά και να δούμε αν πράγματι τέτοια απόβλητα εναποτίθεται εκεί ή όχι. Πιθανότητα είχε κάποιες αποδείξεις ο αναφέρον για να προβεί σε αυτή την αναφορά. Για μια ακόμη φορά θα πρέπει να ζητήσουμε τη γνώμη των ρουμανικών αρχών. Σας ευχαριστώ. Thank you. Uh, first of all, I Ευχαριστώ. Κοιτούσα κάποια έγγραφα πριν από τη συνεδρίαση και από ό,τι φαίνεται ε, ένα από τα δικαστικά όργανα της Ρουμανίας, η δικαστική επιθεώρηση, ε, απέστειλε έκθεση στην οποία αναφέρεται ότι δήθεν ότι μάλλον οι κατηγορίες του αναφέροντος μπορεί να είναι ακριβείς, αυτό που λέει δηλαδή ο αναφέρον μπορεί και να ισχύει ότι κάποιος πήγαινε και να πέθεται ε, ιατρικά απόβλητα σε, κάποιες, ε, σε, κάποιες, σε αυτόν τον χώρο υγειονομικής ταφής και κάποιος άλλος πήγαινε και τα έπαιρνε αυτά τα απόβλητα και τα πολλούσε στην αγορά. Οπότε είναι τελείως διαφορετικά θέματα ε, σε σχέση με τις αναφορές του θέματος 6 όπου το ζήτημα είναι η ρήπανση του αέρα. Διότι αν αυτά που συμβαίνουν, αν πράγματι ισχύουν αυτά που καταγγέλει ο αναφέρον στο σημείο 7, τότε πρέπει να ξεκινήσει ποινική διαδικασία. Οπότε, εγώ θα έλεγα να κρατήσουμε ξεχωριστά αυτά τα δύο θέματα και να την κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά, έω ότου οι ρουμανικέ αρχέ καταφέρουν να καταλήξουν σε ασφαλέ συμπέρασμα για το αν οι κατηγορίε αυτέ ευσταθούν ή όχι. Perfecto. Um, Ωραία έχοντας ακούσει την Κομισιόν και τα μέλη της Επιτροπής, θα ενώσουμε το θέμα αυτό με το σημείο 6. Θα κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή. Στις 18 Σεπτεμβρίου του 2019, ο αναφέρον έστειλε επιστολή όπου αναφέρεται ότι το 2015 η επιχείρηση αυτή κατηγορήθηκε, το 2000, ναι, ναι για διάφορες παρατυπίες μεταξύ αυτών και τη διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων. Αν συμφωνείτε λοιπόν, πέραν της έρευνα που διεξάγει η Κομισιόν, θα πρότεινα να στείλουμε μια... να ζητήσουμε μάλλον από τις Ρωμανικές Αρχές μια επικαιροποίηση της κατάστασης ε, που βρίσκονται όλες αυτές οι ανοιχτές ε, δικαστικές ε, υποθέσεις σε ό,τι αφορά την επιχείρηση αυτή. Οπότε η ΕΠΤΑ θα μείνει ανοιχτή, η Κομισιόν θα συνεχίσει να έρευνα και εμείς ως Κοινοβούλιο θα ζητήσουμε από τις Ρουμανικές Αρχές να μας ενημερώσουν για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι δικαστικές διαδικασίες εναντίον αυτής της εταιρείας. Περνάμε στο σημείο 8, διάφορες αναφορές η 1078 του 2018 ε, της Βελίκα Βελίκοβα, βουλγαρικής ηθαγένειας, φέρουσα 182 υπογραφές σχετικά με την παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου στον ε, οικισμό Τσάρεβετς του Δήμου Μέστρα τη Βουλγαρία. Επίση, άλλη αναφορά με τον αριθμό 1091 του 2018 της Γκαλίνα Τοσέβα, βουλγαρικής ηθαγένεια, με 595 υπογραφέ σχετικά με το αίτημα για τον παροπλισμό τη μονάδα παραγωγή βιομάζας στο Τρούντ τη Βουλγαρίας. Τέλος, η αναφορά 1105 τη Κρεμένα Πέτροβα, βουλγαρική ηθαγένεια, εξ ονόματο της Ένωση η Νόβα Ζαγκόρα θέλει να αναπνεύσει με άλλε 1.176 υπογραφέ σχετικά με τη μονάδα παραγωγή βιαρίου στην Όβα Τζαγκόρα της Βουλγαρίας. Ε, η κυρία Πέτροβα είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθατε. Θα σας δώσω το λόγο για 5 λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ βρίσκομαι εδώ ως εκπρόσωπος της, ε, ε, του συλλόγου μας. Ε, με την ονομασία η Νόβα Ζαγόρα θέλει να αναπνεύσει. Είμαι εδώ διότι τα τελευταία πέντε χρόνια οι βουλγαρικές αρχές δεν επιδεικνύουν καμία επιθυμία να διερευνήσουν τις καταγγελίες που έχουμε κάνει. Πολλοί πολίτες έχουν αναφέρει ε, δυσάρεστες οσμές ε, να ε, προέρχονται από, αυτήν την, από αυτόν την εγκατάσταση βιοαερίου. μόνο φέτος έχουμε λάβει 150 τέτοια μηνύματα. Πολλοί πολίτες υποφέρουν από αυτή την κατάσταση. Στην είσοδο μάλιστα αυτής της εγκατάστασης γίνεται και διαχείριση διαφόρων ειδών ε, ζωικών αποβλήτων ή και άλλων κατηγοριών αποβλήτων που είναι και στερεά και υγρά αλλά που αυτά δεν θεωρούνται απόβλητα βάσει του ορισμού των βουλγαρικών αρχών. Και αυτά τα είδη αποβλήτων μάλιστα εναποτίθενται ε, στην εγκατάσταση αυτή από ε, φάρμες οι οποίες βρίσκονται ε, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Αν, δι, αν μάλιστα συνυπολογίσει κανείς και την ρήπανση του αέρα που προκαλείται εξαιτία αυτή τη εγκατάσταση λόγω τη μεταφορά εκεί όλων αυτών των αποβλήτων με φορτηγά, δεν νομίζω ότι μπορεί κανεί να τη χαρακτηρίσει ω ιδιαίτερα οικολογική αυτή την εγκατάσταση. Το 2017 διαπιστώθηκε ότι δεν είχε γίνει κανένας έλεγχος επί τρία ολόκληρα χρόνια σε υγρά και στερεά απόβλητα που εισέρχονταν στην συγκεκριμένη εγκατάσταση διαχείρισης και τα απόβλητα αυτά μάλιστα αποτίθονταν σε σημείο κοντινό στην ε, εγκατάσταση αυτή και το νερό ε, αποκτούσε μια πολύ δυσάρεστη ε, οσμή, γινόταν καφέ, μύριζε σαν κουτσουλιές, να σας το πω ξεκάθαρα, και δεν ήταν ποτέ σαφές ποια ήταν η αρμόδια αρχή που έπρεπε να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο ζήτημα στη Βουλγαρία. Όταν οικοδομήθηκε, όταν κατασκευάστηκε η συγκεκριμένη εγκατάσταση, επίσης δεν ελήφθη υπόψη η φορά του αέρα στη συγκεκριμένη περιοχή. Κατασκευάστηκε λοιπόν κοντά σε κατοικημένη περιοχή και επειδή το καλοκαίρι ο αέρας, ο άνεμος φυσάει από την εγκατάσταση προς την ε, κατοικημένη περιοχή, προς την πόλη αυτή που βρίσκεται εκεί κοντά, δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα παράθυρά μας. Πολλοί άνθρωποι μάλιστα διαμαρτύρονται ότι έχουν, ότι έχουν ε, ζαλάδες, ότι έχουν πονοκεφάλους και μάλιστα ζητήθηκε και από ανεξάρτητο εργαστήριο να μετρήσει διάφορα είδη αερίων στον, ε, στην ατμόσφαιρα. Τελικά όμως ποτέ δεν έγιναν τέτοιες μετρήσεις. Προσπα... Κανείς δεν προσπαθεί να διερευνήσει τον αντίκτυπο που έχουν αυτές οι δυσάρεστες οσμές στη ζωή των ανθρώπων την καθημερινή. Εμείς πιστεύουμε ότι η μονάδα αυτή βλάπτει την ε, δημόσια υγεία. Γιατί υποφέρουν οι άνθρωποι, λοιπόν. Διότι κατασκευάστηκε η συγκεκριμένη μονάδα με βάση, ορισμένες, ε, με, βάση ορισμένα ψευδή στοιχεία. Δεν είχε ε, εκπονηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Α, και με την ευκαιρία να σας πω ότι καμία μονάδα βιοαερίου στη Βουλγαρία δεν έχει λάβει ποτέ ε, μονάδα περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι κανένας επενδυτής δεν θα ε, ε, έλεγε ποτέ δημοσίως ότι στην πόλη που θα κατασκευαστεί μια, μια τέτοια μονάδα θα αρχίσει να ε, μυρίζει άσχημα ο αέρας. Ε, αυτό που ζητάμε εμεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να καταρτιστούν ορισμένε βέλτιστε πρακτικέ για την καλύτερη διαχείριση και επεξεργασία αυτών των αποβλήπων. Οι πολίτε τη ε, Νόβα Ζαγόρα δεν αντιτίθεται στι πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιθέτω, είμαστε πρόθυμοι να υπερασπιζόμαστε όλα τα περιβλητικά μέτρα που λαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όχι, όχι όταν το αντίτιμο που καλούμαστε να καταβάλουμε είναι η υγεία μας και η υγεία των παιδιών μας. Πρέπει τέτοιου είδους μονάδες να συνοδεύονται από σχετικά μέτρα προστασίας, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει ως οικολογικό το έργο αυτό, την, την μονάδα βιοαερίου αυτή. 20.000 άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να εισπνέουν ε, κακής ποιότητας αέρα και όλε αυτές τις δυσάρεστε οσμές. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Πέτροβα. Τώρα το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. κυρία Αντωνέτα Καλαπής. Thank you, Madam. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω καταρχάς ζητώντας συγγνώμη εκ μέρους των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το γεγονός ότι δεν ε, καταφέραμε να απαντήσουμε και στις τρεις ε, αναφορές. Φαίνεται ότι ε, το ζήτημα αυτό αφορούσε πολλές υπηρεσίες της Κομισιόν και γι' αυτό δεν κατέστη δυνατόν να δώσουμε μια απάντηση. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι είναι πολύ δύσκολο να προσδιορίσουμε την ε, εφαρμοστέα ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι ε, αναφέροντες παραπέμπουν σε διάφορες οδηγίες, αλλά δεν μας δίνουν τη δική τους άποψη για το πώς ακριβώς πρέπει να εφαρμοστούν οι οδηγίες αυτές στην εκάστοτε περίπτωση που αναφέρουν οι αναφορές τους. Τούτων λεχθέντων θα σας δώσω τη δική μας εκτίμηση ανά αναφορά διότι οι αναφορές αυτές βεβαίως αναφέρουν, αναφέρονται σε διαφορετικές ε, εγκαταστάσεις, διαφορετικές μονάδες. Εγώ ε, εργάζομαι στην Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και έχω μαζί μου εδώ τον συνάδελφό μου από τη Γενική Διεύθυνση Καταναλωτών και Υγείας ε, ώστε να τοποθετηθεί και εκείνο αν χρειάζεται. Και μιας και έχουμε μια αναφέρουσα εδώ παρούσα μαζί μας, θα συνεχίσω στα βουλγαρικά. Αναφορά 1078 του 2018. Η αναφορά 1078 του 2018 αφορά την ε, μονάδα παραγωγής ε, βιοαερίου στον οικισμό Τσάρεβετς ε, στο Μέζρα της Βουλγαρίας. Σύμφωνα με τις δημόσιες πληροφορίες που υπάρχουν από, την από τον περιβαλλοντικό έλεγχο που έγινε το 2000, τον Ιούλιο του 2018, έγιναν κάποιοι έλεγχοι λόγω ε, καταγγελιών δυσάρεστων οσμών για δυσάρεστες οσμές που υπήρχαν. Αυτοί οι έλεγχοι, ωστόσο, δεν κατέληξαν στην διαπίστωση συγκεκριμένων παραβιάσεων της νομοθεσίας. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιες ενδείξεις χρήσης ε, διαφόρων υλικών στην μονάδα παραγωγής αυτή που ε, δεν επιτρέπουν την διασπορά αυτών των οσμών, των δυσάρεστων. Έχουν επίσης ληφθεί και άλλα μέτρα και έχουν ε, ακολουθηθεί όλοι οι κανόνες και οι συστάσεις που έχουν δοθεί στη συγκεκριμένη μονάδα. Στη συνέχεια υπήρξαν ε, άλλες καταγγελίες οι οποίες αφορούσαν την ε, ε, απόθεση αποβλήτων βιομάζας. Έγιναν έλεγχοι και τον Φεβρουάριο διαπιστώθηκε ότι τα μη, ε, η μη ρυθμιζόμενη επεξεργασία αποβλήτων συνεχιζόταν. Επομένως, επιβλήθηκε το μέγιστο δυνατό πρόστιμο στη μονάδα παραγωγής βιοαερίου και, στη μονάδα, ε, και στον φορέα που είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά των αποβλήτων και ο ε, φορέας ε, εκμετάλλευσης ε, είναι πλέον υποχρεωμένος να υποβάλει εκθέσεις για την βιομάζα που αποθηκεύεται στη μονάδα του και για την ε, βιομάζα που θα χρησιμοποιηθεί ε, ως λίπασμα. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχουν οι εθνικές αρχές λάβει τα απαραίτητα μέτρα πλέον. Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλαβαίνουν ότι η δυσφορία στους πολίτες είναι πολύ υψηλή, όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, αυτή, δεν, δεν υπάρχει καταρτισμένο πρότυπο για τη μέτρηση, αν θέλετε, των δυσάρεστων οσμών. Αυτό είναι εθνική αρμοδιότητα, οπότε η Κομισιόν δεν δικαιούται να αναλάβει δράση στον τομέα αυτό. Για τις ευρωπαϊκές πράξεις που παρατίθεται στη συγκεκριμένη αναφορά, μπορώ να σας πω τα εξής. Βάσει των πληροφοριών που έχουμε λάβει, εμείς δεν διαπιστώσαμε καμία παραβίαση. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να επαληθεύσουμε μάλιστα και τις πληροφορίες που έχουμε λάβει. Για όλους αυτούς τους λόγους η Κομισιόν δεν θεωρεί ότι χρειάζεται να αναλυφθεί δράση. Αναφορά 1091 του 2018 επίσης. Αυτή η αναφορά αφορά την μονάδα παραγωγής βιομάζας στο Τρούντ της Βουλγαρίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε λάβει, το 2017 ο περιφερειακός ελεγκτής περιβάλλοντος στο Πλόφτιβ έλαβε πολλές καταγγελίες για δυσάρεστες οσμές και θόρυβο που ε, εκπέμπει ε, η συγκεκριμένα μονάδα παραγωγής. Στη συνέχεια έγιναν έλεγχοι, αλλά δεν διαπιστώθηκε κανένας, καμία παραβίαση. Οι αναφέροντες εκφράζουν τι αμφιβολίε του σχετικά με, τους, με τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων. Όμω η Κομισιόν δεν δικαιούται, δεν έχει δικαίωμα να διεξάγει δικέ τη έρευνε, δικού τη ελέγχου για το τι κάνουν ιδιωτικέ εταιρείε προκειμένου να συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και αυτό αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Καταλαβαίνουμε βεβαίως την απογοήτευση των πολιτών ε, της Βουλγαρίας, της συγκεκριμένη περιφέρειας της Βουλγαρίας, όμως πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά ενωσιακά πρότυπα για, το, για τα επίπεδα θορύβου. Αυτό το ζήτημα αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Υπάρχει βεβαίως η οδηγία για τον ε, θόρυβο και δυνάμει αυτής της οδηγίας ε, τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να ε, εκδίδουν χάρτες θορύβου γύρω από αυτοκινητοδρόμους και αεροδρόμια, όμως ε, στην οδηγία αυτή δεν αναφέρονται συγκεκριμένα επίπεδα θορύβου τα οποία θα πρέπει να τηρούνται. Όσον δε τα όσα καταγγέλλονται για μικροσωματίδια στον αέρα και για θόρυβο Υπάρχει μάλιστα μια υπόθεση που εκδικάζεται στο δικαστήριο αυτή τη στιγμή κατά της Βουλγαρίας και μπορώ να σας πω τα εξή. Οι αναφέροντες δεν υποβάλλουν καμία, κανένα αποδεικτικό στοιχείο όσον αφορά την παραβίαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Απλώς παρατίθενται κάποιες ευρωπαϊκές νομικές πράξεις. Ε, για όλου αυτού του λόγου, η Κομισιόν δεν μπορεί να αναλάβει περαιτέρω δράση όσον αφορά την τήρηση τη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η αναφορά 1105 του 2018 αυτό αναφορά το εργοστάσιο αγωγής βιαριού στην Όβα Ζαγόρα της ε, Βουλγαρίας. Αυτό το εργοστάσιο εγκρίθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό 1062. Αυτός ο κανονισμός αφορά την παραγωγή βιοερίου, από διάφορα λιπάσματα κοπριάς. Είχαμε πολλές επιθεωρήσεις γιατί υπήρξαν πολλές καταγγελίες, όμως δεν βρήκαμε να υπάρχουν παραβιάσεις. σε σχέση με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Έτσι λοιπόν μπορώ να αναφέρω τα ίδια επιχειρήματα που προανέφερα. Να πω ότι όταν η κοπριά μετατρέπεται σε βιοαέριο, η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα απόβλητα δεν εφαρμόζεται. Στην περίπτωση αυτή η κοπριά ε, είναι αντικείμενο μεταχείρισης ε, ως ε, προϊόν, παραπροϊόν ζωικό. Έτσι λοιπόν, δεν υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας και γι' αυτό η Κομισιόν σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση δεν σκοπεύει να αναλάβει δράση. Για να συνοψίσω. Να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τους τρεις αναφέροντες. Η παραγωγή βιορίου δεν ε, θα πρέπει να θεωρείται κάτι κακό. Υπάρχουν πολλές καλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν. Όμως όλα αυτά είναι στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και η Κομισιόν δεν έχει κανένα λόγο να παρέμβει. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής μας. Ο κύριος Γκρέφα από το ΕΛΚ μου έχει ζητήσει το λόγο. Για αυτές τις τρεις αναφορές γνωρίζω πολύ καλά προσωπικά τις υποθέσεις. Και τις τρεις. Έχω λοιπόν προσωπική άποψη. Έχω συνεργαστεί με τους ετούντες ε, εδώ και αρκετούς μήνες. Αρκετούς μήνες μάλιστα πριν εκλεγώ μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε μπορώ να σας βεβαιώσω ότι το πρόβλημα είναι πραγματικό είναι πολύ σοβαρό. Η ποιότητα ζωής των κατοίκων αυτών των τριών πόλεων, δύο χωριών και μιας πόλης για την ακρίβεια, ε, κανένα από αυτά δεν είναι μικρό χωριό, ε, η ποιότητα ζωής τους έχει υποβαθμιστεί πολύ. Οι διάφοροι φορείς και τα Ινστιτούτα παραβλέπουν την κατάσταση παρόλο ότι υπάρχουν αναφορές για υψηλές ε, συγκεντρώσεις ε, υδροθείου και αμμονίας επικίνδυνων και δυσάρεστων αερίων. Λέει η Κομισιόν δεν υπάρχουν νομικές, ε, νομική, δεν υπάρχει νομική βάση για τέτοιου είδου ε, καταγγελίες. Αυτό όμως δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται κανεί να είναι ειδικό στη χημεία ή στην ιατρική ή στο περιβάλλον για να καταλαβαίνει ότι η αμμονία είναι ένα τοξικό αέριο και το υδρόθιο επίσης. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι σαφής. Ο, ασφαλής, ε, ο καθαρός και αμόλυντος αέρα είναι δικαίωμα κάθε Ευρωπαίου πολίτη. Το να κρυφτεί κανείς πίσω από γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι μόνο μια πολιτική ομπρέλα και προστασία των επιχειρήσεων που διαχειρίζονται ε, τις μονάδες. Οπότε θα ήθελα να μην είναι ανοιχτέ οι αναφορέ, να ζητήσουμε έκθεση από την Επιτροπή Περιβάλλοντο και μετά ενδεχομένω να επισκεφθούμε και τη Βουλγαρία για να διαπιστώσουμε από κοντά τα γεγονότα. Ευχαριστώ. Perfecto. La señora Maestre. Κύριε Ευχαριστώ πολύ στην ανα... την αναφέρουσα που έκανε ταξίδι και ήρθε εδώ να μας μιλήσει. Ευχαριστώ πολύ την Κομισιόν που μας εξήγησε τη θέση της ακούγοντας και τα δύο μέρη ε, θα συμφωνήσουμε με το ΕΛΚ να μείνει ανοιχτή αναφορά. Ε, λείπουν πληροφορίες. Ε, εμείς τουλάχιστον ως σοσιαλιστές δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα αποτελέσματα των, της έκθεσης ε, της αποστολής και είναι σαφές ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να αναπνέουν ένα καθαρό αέρα. Υπάρχουν λοιπόν θέματα υγείας για τους κατοίκους αυτών των τριών περιοχών οι οποίοι έχουν δικαίωμα να χαίρουν καθαρό αέρα και ψηλό βιωτικό επίπεδο. Ξέρω και άλλες περιπτώσεις μονάδων παραγωγής βιομάζας που δημιουργούν σημαντικές άσχημες σωσμές. Πρέπει και η Βουλγαρία να εξασφαλίσει αυτά τα δικαιώματα που έχουν οι πολίτες της. Άκουσα την... Η κυρία Τόμ, άκουσα την Κομισιόν και μπήκα στη θέση του, της αναφέροντος. Είναι αποκαρδιωτικό να ακούει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν θέλω να στείλουμε αυτό το μήνυμα. Θα ήταν πολύ κακό για την Ευρώπη. Οπότε συμφωνώ να, μείνει ανοιχτή, να μείνουν ανοιχτέ οι αναφορέ και στηρίζω και την πρόταση του ΕΛΚ. Να ζητήσουμε γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντο και να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε λίγο. Γιατί πραγματικά οι άνθρωποι εκεί υποφέρουν και δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, είναι θέμα εθνικό και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ασκήσουμε πίεση. Δίνω το λόγο ξανά στην αναφέρουσα για δύο λεπτά και κλείνουμε έτσι. Έχοντας ακούσει τα μέλη της Επιτροπής μας, ξαναπάρτε παρακαλώ το λόγο. Ναι, ε, είμαι απογοητευμένη από αυτά που άκουσα από την εκπρόσωπο της Κομισιόν. Το γεγονός ότι η εθνική μας νομοθεσία δεν περιλαμβάνει τίποτα για τις κακές οσμές και για το πώς αυτές μετρούνται δεν είναι ικανοποιητικό προφανώς ως απάντηση. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε με τέτοια κακοσμία. Τα δικαιώματά μας προσβάλλονται, κακοποιούνται. Δεν είναι δυνατόν οι νομοθέτες να μας λένε ότι όλα είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αλλά κανείς δεν τολμά να έρθει στα χωριά μας και στις πόλεις μας να μυρίσει τον αέρα. Αν ερχόντουσαν, θα έβλεπαν ότι οι άνθρωποι ξυπνάνε μέσα στη μέση της νύχτας λόγω, των, λόγω της δυσοσμίας. Για φανταστείτε να το είχατε εσείς στο σπίτι σας αυτό. Είναι όρις το πρωί που υποτίθεται θα έπρεπε να ξυπνάμε και να μυρίζουμε φρέσκο ψημένο καφέ. Δεν είναι γεωργικά αυτά τα χωριά, δεν έχουν συνηθίσει τέτοιου είδους οσμές. Ελπίζω ότι θα βρείτε τον κατάλληλο τρόπο για να λύσετε ή να βοηθήσετε να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα, τέτοιου είδου προβλήματα υπάρχουν και σε άλλα κράτη-μέλη. Αυτέ οι μονάδε παραγωγή έχουν παρόμοια προβλήματα παντού. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την αναφέρουσα που βρίσκεται εδώ σήμερα. Αφού ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις κοινοβουλευτικέ ομάδες, αφήνουμε ανοιχτέ τι αναφορέ αυτέ, αλλά ήθελα να πω στην Κομισιόν ότι εμείς θα στείλουμε τις αναφορές το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2000. Στείλαμε τις αναφορές Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2019. Έχει περάσει λοιπόν η προθεσμία ε, βάσει τη οποία ε, θα έπρεπε να μας έχει ενημερώσει η Κομισιόν για την κατάσταση αυτών των αναφορών. Επομένω, ε, ακούσαμε σήμερα την ε, τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όμως ε, θα θέλαμε σας παρακαλέσουμε να μας στείλετε γραπτός όλα τα σχετικά έγγραφα, όλες τις εκθέσεις. Εσείς μας είπατε ότι πήγαν ε, ελεγκτές για να αξιολογήσουν τις αναφορές. Θέλουμε λοιπόν τις αναφορές όλων των επιθεωρηθών που αξιολόγησαν την κατάσταση και τις φερόμενες παραβιάσεις. Επίσης, θα ζητούσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας γνωστοποιήσει το εξή Εσείς ε, έχετε προσφύγει κατά του κράτους μέλους, γιατί δεν ε, μας το εξηγήσατε. Ε, έχετε απευθυνθεί στο κράτος μέλος, έχετε απευθύνει κάποια προσφύγη κατά του κράτους μέλους και αυτό να μας το στείλετε γραπτός. Και επίση, εμεί, από την πλευρά τη Επιτροπή Αναφορών θα στείλουμε στη μόνιμη αντιπροσωπεία τη Βουλγαρίας έτοιμα να μα ενημερώσει για αυτέ τι αναφορέ που έχει λάβει Επίσης ε, θα τις κοινοποιήσουμε τις ανησυχίες της Επιτροπής μας και θα ζητήσουμε τις βουλγαρικές αρχές να προβούν ε, στις ε, κατάλληλες εκτιμήσεις επιπτώσεων. Όμως, να μας ενημερώσει η Κομισιόν τις εξυλογήσεις που έκανε το κράτος μέλος, που και εσείς αξιολογείτε με τους δικούς σας επιθεωρητές στις αξιολογείτε τις εκθέσεις του κράτους μέλους, θα θέλαμε να τις διαβιβάσετε αυτές στην Επιτροπή μας. Επίσης, δεχόμαστε την ε, πρόταση του ΕΛΚ να σταλεί μια γνωμοδότηση, ναι, συγγνώμη, να σταλεί έτοιμα γνωμοδότηση και στην ΕΝΒΗ και κάποιο μέλος του ΕΛΚ ζήτησε μια πιθανή αποστολή να μεταβεί στη Βουλγαρία για να επισκεφτεί αυτούς τους ε, δήμους Ακριβώς ε, πριν λίγο εγκρίναμε τις αποστολές και να πω στους συντονιστές ότι για το δεύτερο εξάμεινο του 2020 θα μπορούσατε να αιτηθείτε αυτής της αποστολής που ζήτησε το ΕΛΚ. Αφήνουμε ανοιχτέ λοιπόν αυτές τις αναφορές. Η Επιτροπή θα στείλει στη μόνιμη την προσωπία της Βουλγαρίας ε, όλες τις αναφορές για να μας απαντήσει τη θέση του κράτους μέλους και απαιτούμε από την Κομισιόν να μας στείλει όλες τις εκθέσεις που έχουν υλοποιηθεί. Sí, να μας ενημερώσει αν έχετε προσφύγει κατά του κράτους μέλους και να αξιολογήσετε τις εκθέσεις του κράτους μέλους. Para que Θα στείλουμε και στην ΕΜΒΙ έτοιμα για γνωμοδότηση και οι συντονιστές θα ζητήσουν την υλοποίηση αποστολής στη Βουλγαρία. Αν συμφωνείτε όλοι, Αυτές είναι οι αποφάσεις που λάβαμε εδώ για αυτές τις αναφορές. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν την αναφέρουσα, την κυρία Πέτροβα, που παρευρέθη εδώ σήμερα. Να περάσουμε τώρα στην επόμενη αναφορά, στο σημείο 9 της Μερσής διάταξης, 1099 του 2018 του Ιώζεφ Στρασκόφσκι, από την Πολωνία ενδιαφέρουσα 531 υπογραφές σχετικά με την περιοδική καταστροφή που προκαλείται από το υπεύθυνο σαρκορυχείο στην Ανατολική Πολωνία. Δεν βρίσκεται εδώ το ο αναφέρον, επομένως να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο κύριο, στον κύριο Μπλόντα Βάρισικ. Σας ευχαριστούμε. Uh, thank you very much, Madam Ευχαριστώ, Πρόεδρε. τον Οκτώβριο του 2008 οι υπηρεσίες της Κομισιόν έλαβαν μια καταγγελία σε ό,τι αφορά πιθανές αρνητικές επιπτώσεις σε δύο τοποθεσίες που προστατεύονται από τις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους που προκαλείται από το υπαίθρο αρχείο εξόριξη στο Μισλάβιτς. Βρίσκεται η τοποθεσία 7 χιλιόμετρα από δύο περιοχές Natura 2000. Η μία είναι μια ειδική περιοχή προστασίας, η να στο πράσικα και η λίμνη Γκλόπμου. Τα χαρακτηριστικά και των δύο τοποθεσιών ε, σχετίζονται με την προστασία υγροβιοτοπών και φυσικά αυτό εξαρτάται από τις ε, συνθήκες της λίμνης Γκόπλο. Αυτές οι ε, εξορρυκτικές διαδικασίες οδηγούν στη μείωση του επίπεδου των υπογείων υδάτων ε, επειδή χρησιμοποιούνται ε, τα ύδατα στο ορυχείο. Η Κομισιόν έστειλε ε, μία πρώτερη αποστολή για τις επιπτώσεις του άρθρου 6264 σε σχέση και με το άρθρο 7 της Οδηγίας για τους οικοτόπους. Στην απάντηση της αιτιολογημένης γνώμης, η Πολωνία αναφέρθηκε στα απορίσματα του αριθμητικού και ιδρυολογικού μολέντου ε, ένας υπάρχει ένας διευρυμένος κόνος καταπτώσης που έχει δημιουργηθεί από το ρηχείο και δεν επηρεάζει τους προστατευόμενους οικοτόπους και τα ενδύματα των ειδών στις περιοχές του δικτύου Natura 2000. Επίσης, ε, τα αποτελέσματα της παρακολούθησης ε, των οικοτόπων μας έδειξαν ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές ε, στις σχέσεις στην περιοχή της λίμνης Γκόλπος ό,τι αφορά τα ύδατα. Ούτε μας έδειξαν επιδείνωση των ενδιατημάτων και των οικοτόπων. Οι εξηγήσει που δόθηκαν από τις πολωνικές αρχές κρίθηκαν επαρκείς από την Κομισιόν και σε αυτή τη βάση η Επιτροπή σταμάτησε, έκλεισε τη διαδικασία επί παραβάση στις 11 Απριλίου 2019. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τα μέλη, παρακαλώ κυρία Άουκεν. Κοιτάξτε, έχω λίγο εκπλαγή που Είχαμε ισχυρισμού παραβιάσεων και κατόπιν ακούσαμε τη σχολή τη Κομισιόν ότι όλα πάνε καλά. Τι μα λέει η Κομισιόν, όλα είναι τέλεια. Επειδή η πολωνική κυβέρνηση είπε ότι όλα είναι καλά. Και δεν έχουμε εδώ του αναφέροντες. Ούτε έχουμε την απάντηση. Θα ήθελα να είμαστε δίκαιοι εδώ. γιατί έχουμε και την ε, περίπτωση της Γαλλικίας με τα ορυχεία και έχουμε παρόμοια προβλήματα σε πάρα πολλές τοποθεσίες. Η μόνη απάντηση είναι της πολιτικής κυβέρνησης που λέει ότι δεν υπάρχει αντίκτυπος στο δίκτυο Natura 2000. Ωραία. Είδα και την ισπανική απάντηση από τη Γαλλικία χθε το βράδυ στα ισπανικά. Τα διάβασα, δεν ήταν και εύκολο και εκεί μα έλεγαν όλα πάνε πολύ καλά. Και έχω μπορώ να σα πω ότι δεν είναι. Να δώσουμε μια ακόμη ευκαιρία λοιπόν σα ζητώ και να δώσουμε τη δυνατότητα στον αναφέροντα να απαντήσει και να δούμε αν μπορούμε να δώσουμε συνέχεια. Ναι, θέλω απλώς να επαναλάβω αυτό που είπε και η συνάδελφος κυρία Άουκεν. Το πρόβλημα είναι συστημικό και με εκπλήσει και μένα ε, ιδιαίτερος η απάντηση που ακούσαμε από την ε, Κομισιόν γιατί η εξόριξη λιγνίτη είναι πρόβλημα. Εμείς ως Επιτροπή Αναφορών έχουμε λάβει και αναφορά από την Ανατολική Γερμανία στο τέλος της τελευταίας κοινοβουλευτικής θετίας και είχαμε ε, πραγματοποιήσει και μια ερευνητική επίσκεψη στην ε, Σαξονία της Ανατολικής Γερμανίας και είδαμε με τα μάτια μας ε, πόσο σοβαρές ε, και αρνητικές είναι οι επιπτώσεις στη φύση από αυτήν την εξορρυκτική δραστηριότητα και τα συμπεράσματα τα οποία καταλήξαμε ήταν επίσης πάρα πολύ αρνητικά. Οπότε θα παρακαλούσα και εγώ να μην κλείσει η αναφορά αυτή και να ακούσουμε σε πρώτη φάση τουλάχιστον και τις απαντήσεις του αναφέροντος ε, στα όσα ακούσαμε από την Επιτροπή. Κυρία Τόμ. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να επαναλάβω. Απλώς να πω ότι ακούσαμε πριν μισή ώρα την αναφορά για τα ιατρικά απόβλητα και εκεί ακούσαμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και εκεί ο συνάδελφός μας ήταν ε, που μας είπε ότι έλαβε έκθεση και ότι αυτό από μόνο του αποτελεί απόδειξη ότι δεν συμβαίνει τίποτα κακό. Ε, όχι, δεν είναι έτσι. Πρέπει να μείνει η αναφορά ανοιχτή, ώστε να μπορέσει και ο αναφέρον να αποδείξει ότι αυτά που ε, ισχυρίζεται ευσταθούν. Yeah, thank you. Ο κ. Κροσνοντεύσκη, να ευχαριστώ πολύ. Σε αντίθεση με πολλούς συναδέλφους, εγώ ξέρω την περιοχή, γιατί έχω εκλεγεί στην περιοχή αυτή, την έχω επισκεφτεί και έχω και κάποια εμπειρογνωμοσύνη. Δεν είναι λοιπόν ξεκάθαρη η κατάσταση. Γενικά θα έλεγα εντυπωσιάστηκα πως καλλιέργησαν εκ νέου αυτή την περιοχή. και θα ξέρετε ότι το 2030 θα κλείσουν τα ορυχεία γενικώ στην Πολωνία. Όμως νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά αυτές τις ανησυχίες ε, των πολιτών. Η δική μου ομάδα πρότεινε στην Επιτροπή Βιομηχανίας ε, να υλοποιήσει μια αποστολή στην περιοχή αυτή και αν κάποιο από τη δική σας Επιτροπή θα ήθελε να συμμετέχει, αν εγκριθεί η αποστολή βεβαίως, θα το εκτιμούσαμε και εγώ προσωπικά. θα έλεγα ότι ίσως δεν είναι τόσο δραματική η κατάσταση όπως περιγράφεται ίσως στην αναφορά, αλλά φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το τι λένε οι πολίτες και ποιες είναι οι ενισχύες τους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, κάνεις Θα προσπαθήσω να σας τα πω πολύ σύντομα. Κάποιες αναφορές πρέπει κάποιες στιγμές να κλείνουν. Δεν μπορούμε να κρατάμε όλες τις αναφορές ε, ανοιχτές. Εν τούτης, θεωρώ ότι δεν είναι η στιγμή να κλείσουμε αυτήν την συγκεκριμένη αναφορά. Πρέπει να την κρατήσουμε ανοιχτή. Και πέραν των επιχειρημάτων που ακούστηκαν ήδη, νομίζω ότι το ζήτημα των ανοιχτών ε, λιγνητορυχίων στην Πολωνία και όχι μόνο στην Πολωνία είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα έτσι και αλλιώς. Και νομίζω ότι υπάρχει και μια αντίφαση ε, ανάμεσα στην, ε, μια αντίθεση αν θέλετε, ανάμεσα στην ε, ανοιχτή εξόριξη λιγνίτη και στη γεωργία. Εγώ έχω συνομιλήσει και με Πολωνούς συναδέλφους για το ζήτημα αυτό και καταλαβαίνω ότι βρίσκει βρίσκονται σε εξέλιξη και κάποιε διαδικασίε τροποποίηση τη ισχύουσα νομοθεσία στην Πολωνία. Οπότε θα πρέπει να, να ολοκληρωθούν πρώτα αυτέ τι διαδικασίε, να δούμε αν θα λυθεί το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο και αν πράγματι γίνει και ερευνητική αποστολή από άλλη επιτροπή, ενδεχομένω θα ήταν ε, σωστό να συμμετάσχουν μέλη και τη δική μα επιτροπή, προκειμένου να διαπιστώσουν και οι δύο ισόμαστε τι συμβαίνει εκεί. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μέστρε, ευχαριστώ. Επίσης να πω ότι δεν μπόρεσαν να έρθουν αναφέροντε ε, και καθώς έχουμε μόνο τη μία εκδοχή τη πολεμική κυβέρνηση. εγώ συμφωνώ με την πλειοψηφία των βουλευτών στο ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Και αν είχαμε και τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στην αποστολή τη Ήτρα θα ήταν ιδανικό. Να βρούμε μια συμφωνία με τον βουλευτή ή με την ε, ομάδα που θα υλοποιήσει αυτή την επιστολή. Θα ήταν ευκαιρία για να διαρευνήσουμε περισσότερο το θέμα. Αλλά πάμε είτε όχι στην αποστολή να διατηρήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά για να εξετάζουμε περισσότερο εις βάθος το ζήτημα. Ευχαριστώ. Κυρία Άουκεν εκ νέου. Κοιτάξτε, εγώ ήμουν σε αυτή την αντιπροσωπεία πέρσι στη Σαξονία και είχαμε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα από την μόλυνση από τα ορυχεία. Είχαμε πολύ βαριά μόλυνση. Και φυσικά, οι πάλι οι αρχές έλεγαν ε, δεν τρέχει τίποτα. Εγώ σέβομαι απόλυτα ανθρώπους που έχουν εκλεγεί στην περιοχή αυτή. Θα ε, υπάρχουν διλήμματα όμως, αλλά πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε αυτά και να λέμε. Όλα είναι εντάξει, γιατί δεν είναι εντάξει αυτή η διαδικασία εξορίξεων, επιδεινώνει το κλίμα αλλά ε, μάλλον ε, ο Λιγνίτης ε, και ο Άνθρακας συνεισφέρουν πολύ περισσότερο στην επιδείνωση του κλίματος. Όμως είναι σημαντικό να επισκεπτόμαστε και αυτές τις περιοχές. Just... Uh, Θα ήθελα να τονίσω είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο να συγκρίνουμε τη Σαξονία με αυτή την περιοχή. Με το χάρη είχαμε ένα μεγάλο λιγνητικό εργοστάσιο που παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έκλεισε πρόσφατα. Και επίσης ε, σιγά σιγά θα κλείνουν ε, και τα ορυχεία στο μέλλον. Και αυτό είναι ιδιαίτερα επίμαχο. Γιατί όταν μιλάς ε, με τον κόσμο εκεί, με τους πολίτες, υπάρχουν το θέματα της ανεργίας, ξέρετε όλα αυτά που δείχνουν ακόμη περισσότερο πόσο σημαντικό είναι το τι τονίζουμε και σε άλλες επιτροπές, δηλαδή η δίκαιη μετάβαση και το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση. Έτσι λοιπόν, δράτω την ευκαιρία για να απευθύνω έκκληση για να το υποστηρίξετε αυτό και στο μέλλον, στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εγώ θα υποστηρίξω ότι θα στείλουμε το λογαριασμό στα εγγόνια μας, όπως προτείνετε τώρα. Λοιπόν, αφού ακούσαμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες, να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή. Η πρόταση θα ήταν... Καταρχήν, να στείλουμε μια επιστολή στην Επιτροπή Βιομηχανίας, αν εγκριθεί η αποστολή της ΣΥτΡΕ, ότι θα θέλαμε και εμείς να συμμετέχουμε με ένα-δύο μέλη της Επιτροπής μας στην αποστολή αυτή. Η δεύτερη πρόταση είναι να στείλουμε επιστολή στην πολωνική κυβέρνηση για να τους εξηγήσουμε ότι η Επιτροπή Αναφορών ανησυχεί για το περιβαλλοντικό αντίκτυπο και για το ότι δεν έχει γίνει νέα αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ζητάμε επικαιροποίηση της κατάστασης. Και αν συμφωνείτε να στείλουμε και επιστολή στον αναφέροντα εξηγώντα του ποια είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να μας γνωστοποιήσει αν θέλει να διατηρηθεί ανοιχτή αυτή η αναφορά. Συμφωνείτε? Αν συμφωνείτε, συμφωνούμε σε αυτά. Και να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης, υπαριθμόν 10, η αναφορά 0059-2017 του Ισμαήλ Αντώνιο Λόπες Πέρες, Ισπανικής Ιθαγένειας, εξ ονόματος ε, της ε, Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Ένωσης Πετών Ντολόμπο, σε σχέση με το ρηχείο Βολφραμίου στο Λουσάν της Γαλλικίας βρίσκεται εδώ ο αναφέρον, ο Ιωάν Εύαν Σπιν. Θα του δώσω καταρχήν, θα τον καλωσορίσω στην ε, Επιτροπή μας και θα του δώσω το λόγο για πέντε λεπτά για να μας παρουσιάσει το θέμα. Καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας μιλήσω. Ήθελα να σας ενημερώσω για τις ε, βασικές παραβιάσεις του, του ευρωπαϊκού δικαίου σε ό,τι αφορά την ε, πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, περιβαλλοντικές μελέτες, διαχείριση των αποβλήτων σε ε, διαδικασίες εξόριξης στη Γαλλικία. Οι υδρολόγοι έκαναν μια επιθεώρηση, ο κύριος Στίβεν Έλμερμαν συγκεκριμένα, ειδικό, που επισκέφθηκε αυτή την περιοχή, καθώς επίσης και άλλες περιοχές κοντά στο Σαντιάγο. Ο Δόκτωρ Έμερμαν μας ενημέρωσε ότι υπάρχουν σαφή, ε, σαφείς ενδείξεις εσωτερικής υγροποίησης. Βλέπετε στη φωτογραφία. Το ίδιο έχει γίνει στην Ιταλία, στην Ρουμανία, στη Βραζιλία και σε άλλες περιοχές της Ισπανίας. Ο Γενικός Διευθυντής ε, Ορυχείων της Γαλλικίας ήδη ελέγχεται για περιβαλλοντικά εγκλήματα ε, σε ορυχεία και καμιά ντουζίνα περίπου περιο... αντίστοιχα ορυχεία της ε, Γαλλικίας βρίσκονται επίσης στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών. Η γαλλικιανή κυβέρνηση πολύ, σύντο, πολύ πρόσφατα μας έστειλε απάντηση ε, αναφέροντας ε, τα συμπεράσματα του επιθεωρητή, ο οποίος έλεγξε την περίπτωση. Λέει η απάντηση αυτή ότι ε, τα φράγματα χτίστηκαν για λόγους παραγωγής υδροελεκτρικής ενέργειας και συνεπώς θα πρέπει Ε, το θέμα να το αναλάβει, να το διευκρινίσει η υδρολογική υπηρεσία παρόλο που ε, στα φράγματα ε, συλλέγονται, ε, αποτίθενται υλικά ορυχείων. Να σας δώσω μια, ένα παράδειγμα για να δείτε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Τα μεγαλύτερα, αυτό το μεγάλο φράγμα χτίστηκε το 1939 από μια Βρετανική εταιρεία, θα δείτε ότι το 1940 υπάρχει μια έκθεση για το πώς χτίστηκε το φράγμα αυτό στην σελίδα 10 της έκθεσης που βάλαμε πέρσι στην Επιτροπή. Ε, το 1960 το φράγμα αυτό έσπασε και δημιούργησε, προκάλεσε μια σημαντική καταστροφή. Υπάρχει κι άλλο ένα μικρότερο. Τα δύο αυτά εμφανίζονται μέχρι το 2000 σε, όλα τα, σε όλες τις αιτήσεις εκθέσεις ε, για τα ορυχεία. Βλέπετε τα προγράμματα εργασίας του ορυχείου από το 1966, 1996 μέχρι το 2000 και βλέπετε ότι εμφανίζονται τα φράγματα αυτά. Επίσης συμπεριλαμβάνονται ε, στην καταγραφή ε, των φραγμάτων που σχετίζονται με ορυχία στην Γαλλικία. Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, λέμε. Έτσι είναι και αυτή η περίπτωση. Όλα τα τοπικά έγγραφα, μάλλον σε κανένα τοπικό έγγραφο δεν αναφέρεται ότι αυτά τα φράγματα χτίστηκαν για παραγωγή υδροελεκτρικής ενέργειας. Προφανώς η απάντηση της Γαλλικίας αποτελεί κοροϊδία σε ό,τι αφορά το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακόμα και η ίδια η εταιρεία του ορυχείου ε, έχει εκθέσεις ανησυχητικές σε ό,τι αφορά την μόλυνση των υδάτων. Δεν έχει γίνει μελέτη περιβαλλοντικής ε, ε, εκτίμησης και η εγκατάλειψη του ορυχείου δείχνει έλλειψη, πραγματική συστηματική έλλειψη ελέγχου συστηματικά παραβιάζονται οι ευρωπαϊκές οδηγίες και οι νόμοι που τις μετέγραψαν στην Ισπανία. Η γαλλικιανή κυβέρνηση εξακολουθεί να παρεμποδίζει τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες. Ζητούμε να έρθετε επιτόπου για να διαπιστώσετε η διεισόμαση της παραβιάσης αυτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης θα πρέπει να επιτελέσει το καθήκον της να παρακολουθεί την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον κύριο Φερνάντες Γκόμες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην περίπτωση αυτή, η Κομισιόν ε, έχει ενώπιον της μία αναφορά, όπου υπάρχει καταγγελία για τον ε, περιβαλλοντικό αντίκτυπο της περιβαλλοντικής επιπτώσεις ε, ενός ορυχείου βολφρεμίου όπου δεν έχουν ε, γίνει σεβαστές οι υποχρεώσεις της οδηγίας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στην πρώτη αξιολόγηση που έγινε από την Κομισιόν εξήχθη το συμπέρασμα ότι δεν μπορούσε να διαπιστωθεί κάποια παραβίαση της οδηγίας βάσει του ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες μας έδειχναν ότι στην πραγματικότητα δεν επρόκειτο για μία νέα άδεια, αλλά απλώς για αλλαγή του κατόχου. Ωστόσο, η Κομισιόν εξέτασε τις νέες πληροφορίες που μας ε, διαβίβασαν οι αναφέροντες και εκ νέου δεν βρήκε κάποια ένδειξη παραβίασης της οδηγίας. Στην περίπτωση αυτή, η Κομισιόν επίσης παρέμπεψε στην ανακοίνωση της Κομισιόν που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2017 σε σχέση με την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης όπου γίνεται πιο στρατηγική εστίαση για τη θέσπιση κριτηρίων σχετικά με τις ε, προτεραιότητες ε, των ε, ε, δράσεων που υλοποιεί η Κομισιόν για την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Στην ανακοίνωση αυτή προβλέπεται ότι με μονομένες περιπτώσεις μη ορθής εφαρμογής που δεν επιτρέπουν να αξιολογήσουμε ευρύτερα ζητήματα δηλαδή που να δημιουργούν ε, ένα συστημικό πρόβλημα κακή εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, ε, θα πρέπει να κρίνονται από τα αρμόδια δικαστήρια, γιατί αυτά διαθέτουν ε, τα κατάλληλα και πιο επαρκή μέσα για να αξιολογήσουν τα ζητήματα αυτά. Επομένως, η Κομισιόν παρέπεμψε τους αναφέροντες στο να χρησιμοποιήσουν αυτά τα ένδικα μέσα σε εθνικό επίπεδο για να καθοριστεί αν ε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε σχέση με την εφαρμογή των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ε, νομοθεσία της Ένωσης και που αποτελούν φυσικά και μέρος του εθνικού δικαίου εφόσον έχουν ε, μεταφερθεί στο ισπανικό δίκαιο. Σας ευχαριστώ. Τελειώσατε. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τώρα στις παρεμβάσεις των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Μέστρα. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι κατά την έποψή μας, πού να το πιάσουμε αυτό το θέμα. Γιατί δεν ε, είναι μόνο ότι είναι θολή η διαδικασία, γιατί είναι σουμπιούντιτσε, η διαδικασία, δηλαδή κρίνεται για πιθανά περιβαλλοντικά εγκλήματα, αλλά βάσει και των ε, στοιχείων βλέπουμε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μόλυνσης ή υπάρχει πραγματική μόλυνση. Και κοιτάξτε, μας εκπλήσει που πρέπει να δούμε σήμερα να έρχεται ακριβώς μία έκθεση, ενώ μας λέει εδώ και ένα χρόνο αναφέροντας ότι περιμένει ε, απάντηση από την κυβέρνηση της Γαλλικίας για το θέμα αυτό. Και η τηλόγηση ναι, είναι ότι η οδηγία περιβαλλοντικού αντικτύπου ε, ή στον ε, νόμο της περιφέρειας υπάρχει μία διάταξη ότι, που λέει ότι η εγκατάσταση είναι από το 39 ε, και επομένως δεν μπορεί να εφαρμοστεί η νομοθεσία, αυτό προκαλεί ανασφάλεια στους πολίτες. Δηλαδή δεν στέκει αυτή η αιτιολόγηση. Εμείς φυσικά πετούμε να είναι ανοιχτή αναφορά και να πετηθεί από την κυβέρνηση της Γαλλικίας να ληφθούν ε, οι απαραίτητες δράσεις για να σταματήσει η λειτουργία της εγκατάστασης αυτής επίσης η Ερμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος να ε, προβεί σε κατάρτιση γνωμοδότησης. Θα ήταν καλό να επισκεφτούμε και την τοποθεσία για να, να γνωρίσουμε καλύτερα την υπόθεση. Γιατί ε, εδώ μας δίνουν κάποιες ε, εκθέσεις για να μας βοηθήσουν να, να μας γνωστοποιήσουν τα πράγματα, αλλά μας τις δίνουν καθυστερημένα. Έτσι λοιπόν, είδαμε κάποιους φακέλους όπου παρουσιάζονται οι επιπτώσεις, είδαμε και τις φωτογραφίες του αναφέροντα όμως ότι ήταν καλύτερα να πάμε εκεί επιτόπου και να συνομιλήσουμε και με τους εμπειρογνώμονες. Ευχαριστώ κύριε Άουκεν. Είμαι σοκαρισμένη από αυτά που είπε η Κομισιόν. Όχι εσάς προσωπικά, έτσι. Αλλά ακούσαμε τον Επίτροπο Σεύκοβιτς Τη προάλλη να λέει είναι μια ε, μεμονωμένη περίπτωση, δεν χρειάζεται να λάβουμε υπόψη. Ε, θα ζητήσουμε να γίνει εκ των υστέρων υπερβολοντική μελέτη. Τι θα πει εκ των υστέρων. Εκ των υστέρων σημαίνει κατόπιν εορτής, ε, αφού έχουν πεθάνει οι άνθρωποι. Τι, τι λέει τώρα η Κομισιόν, ότι οι μεμονωμένοι αναφέροντες δεν αξίζουν προσοχής ακόμα και αν γίνεται παραβίαση του, της, της ε, ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Και δεν είναι και μόνο την περίπτωση. Είναι συστημικό το πρόβλημα. Το, έχουμε, το ακούμε στη Γαλλική εδώ και πολύ καιρό. Προφανώς είναι προσβλητικό να μας στέλνουν μετά από ένα χρόνο επιστολή χτες στα Ισπανικά. χωρίς να προλάβουμε ούτε να τη μεταφράσουμε. Και να μας λένε μάλιστα ότι και όλα είναι εντάξει. Σίγουρα πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά και να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να πούμε στην Κομισιόν ότι ένα από τα πιο βασικά της καθήκοντα είναι θεματοφύλακα της συνθήκης. Is this back? sorry. sorry, sorry. Ζητώ συγγνώμη που χτυπάει το κινητό μου τηλέφωνο. Κοιτάξτε τι είπε ο, ο Πίτροπος Σεύκοβιτς τις προάλλες. Ότι αν είσαι μεμονωμένος δεν σε παίρνουν στα σοβαρά. Όχι Κομισιόν. Θέλουμε να επιτελέσετε το καθήκον σας του θεματοφύλακα των συνθήκων. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε μέχρι όλα να γενικευτούν. Το επιχείρημα το ότι πρόκειται για παλιό ρηχείο δεν χρειάζεται, ε, επειδή είναι παλιό ρηχείο δεν χρειάζεται καινούργια περιβαλλοντική μελέτη, δεν ισχύει. Και μετά οι υπερβαλλοντολόγοι, οι οικολόγοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες. Και έχουμε και την οδηγία για την ποιότητα των υδάτων που παραβιάζεται. Και τι λέτε τώρα, όλα να γίνουν εκ των υστέρων, τα θάνατον δηλαδή. Και στη Βιέννη είχαμε παρόμοια προβλήματα και τα καταφέραμε. Σας παρακαλώ πολύ, Κομισιόν, Κάντε το καθήκον σας. Χαίρομαι και για τη στάση του ΕΛΚ, να σας πω την αλήθεια. Γιατί μετά το, το θέμα των οσμών που κοιτούσαμε προηγουμένως, ε, έχουμε αυτό το, αυτή τη θετική στάση. Χαίρομαι. Muchísimas gracias, señora Ευχαριστώ. Ε, πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ακούσω κάποια περαιτέρω σχόλια από την Κομισιόν. Γιατί δεν επιμείνατε να λάβετε έγκαιρα τις απαντήσεις από τις αρχές της Γαλλικίας. Είναι πολύ περίεργο το γεγονός ότι λάβαμε τις απαντήσεις αυτές ε, τελευταία στιγμή στην πραγματικότητα. Εσείς ευθύνεστε γι' αυτό. Όπως και να έχει πάντω είναι απαράδεκτο. Αυτό δεν είναι τρόπος εργασίας. Δεν είναι δυνατόν για έναν ολόκληρο χρόνο να μην έχουμε απαντήσεις. Και αν ευθύνονται κατά κύριο λόγο οι αρχέ Γαλλικία, φταίτε και εσείς όμως, που δεν επιμείνατε να τι λάβετε νωρίτερα τι απαντήσει. Όσον αφορά την ε, επίσκεψη που έγινε πριν από 10 χρόνια στην Γαλλικία με ε, αντικείμενο την ε, μόλυνση του ποταμού του Ρίας. Και εκεί ήταν σαφές ότι υπήρχε σοβαρότατη μόλυνση και ενώ συνέβαιναν αυτά μπροστά μας, οι αρχές μας έλεγαν όχι, όχι, όλα μια χαρά είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και παρά το γεγονός ότι εμείς καταλήξαμε τότε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα, οι αρχές μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει λόγος να φιλτραριστεί το νερό. Τώρα τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Γιατί στην ίδια περιοχή ε, τελικά ε, βλέπουμε εδώ ότι ε, παράγονται και τρόφιμα. Έχουμε δηλαδή τα, τα προϋπάρχοντα προβλήματα τα περιβαλλοντικά τώρα έρχονται να προσθεθούν σε αυτά τα προβλήματα και τα προβλήματα από την εξορρυκτική δραστηριότητα. Είναι απαράδεκτο να γίνεται κάτι τέτοιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην αναλαμβάνει κανεί δράση. Οπότε θέλω να ευχαριστήσω καταρχά τον αναφέροντα για το γεγονό ότι έθεσε το θέμα. Και ενστερνίζομαι κι εγώ, υποστηρίζω κι εγώ την ε, πρόταση, όχι μόνο να μην είναι ανοιχτή η συγκεκριμένη αναφορά, αλλά να κάνουμε και μια ε, ερευνητική επίσκεψη γιατί εμπλέκονται πάρα πάρα πολλοί ε, άνθρωποι και φορείς ε, στην παραγωγή τροφίμων. Ευχαριστώ κύριε Ροδρίγης. Muchas gracias, Presidenta. Ε, Ευχαριστώ. Στην Επιτροπή αυτή παρευρίσκομαι για να υποστηρίξω την, το αίτημα του αναφέροντος. Ήδη το έκανε η ομάδα μου όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η καταγγελία σε αυτή την επιτροπή από την Ένωση Πετών Ντολόμπο όπου ακριβώς ε, αναφερόταν στην επανέναρξη μιας εξορρυκτικής δραστηριότητας. Ε, πρόκειται για ένα ρηχείο που είχε σταματήσει τη δραστηριότητά του στα τέλη του 19ου αιώνα και είχε δοθεί η νέα έγκριση για να ξεκινήσει τις δραστηριότητε τους και να χρησιμοποιήσει κάποιες εγκαταστάσεις που είχαν ε, φτιαχτεί το 1939 χωρίς ε, να υπάρχουν οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσει ε, για να μπορούν να κρατήσουν ουσιαστικά τα πόβλητα της νέας εξορρυκτικής δραστηριότητα. Δεν έγινε καμία μελέτη επιπτώσεων, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ούτε λήφθησαν υπόψη οι ενδιαφερόμενοι. Ε, αν ε, είχε γίνει η ακρόση, θα ε, γίνονταν εμφανείς και οι κίνδυνοι που ενέχονται υπήρξαν ε, σοβαρές ενδείξεις ε, ότι μπορεί να πληγεί πολύ σοβαρά η υγεία των ατόπων εφόσον δεν πληρούνται οι ελάχιστες τεχνικές ε, προϋποθέσεις αυτών των δεξαμενών για να μπορέσουν να κρατήσουν τα λύματα. Εκεί υπάρχουν σοβαρά σοβαρή κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, γιατί έχουμε βαρέα μέταλλα κτλ. Επίσης υπάρχει μεγάλο κίνδυνο για την βιοπικιλότητα της περιοχής. Ε, ε, από εκεί περνά ο ποταμό ε, Φίνς και μπορεί να προκαλέσει να προκληθούν πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην βιοπικιλότητα και στα είδη της περιοχής αλλά και πολύ μεγάλες επιπτώσεις για όλη την περιοχή και μπορεί να έχει υπάρξει κοινωνικός ε, και εργασιακός αντίκτυπος. Μπορεί να πληγεί η καλλιέργεια των ε, μαλακίων, ε, καθώς πάρα πολλές οικογένειες δραστηριοποιούνται στην περιοχή σε αυτή τη δραστηριότητα και καθώς ε, δεν υπάρχουν ε, οι απαραίτητες ε, υγειονομικές προϋποθέσεις μπορούμε να έχουμε σοβαρές επιπτώσεις. Υποστηρίζω λοιπόν τον αναφέροντα και ζητώ από την Επιτροπή να διατηρηθεί ανοιχτή η αναφορά. Και από τότε που κατατέθηκε η αναφορά μέχρι σήμερα υπάρχουν κάποια στοιχεία που θα πρέπει να μας οδηγήσουν στο να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Η εισαγγελία έχει ε, απαγγείλει μάλιστα και κατηγορίες στον Γενικό Διευθυντή Ορυχείων και Ενέργειας για εγκλήματα που έχουν να κάνουν ακριβώς ε, με τις αιτίε ε, που διέπουν αυτή την αναφορά. Δηλαδή, ε, παίρνοντα χάρη αβάθμιση του περιβάλλοντο που προκύπτει από το νέο άνοιγμα του εργείου χωρί να υπάρχει περιβαλλοντική μελέτη. Επίση, ε, ε, αποδίδει ευθύνε λόγω των της κατάστασης στην οποία βρίσκονται αυτές οι δεξαμενές και πρέπει να αναφέρω και κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή την Επιτροπή. Έχει ζητήσει να αναφέρει στο αν έχουν συμμετέχει ή ενδιαφερόμενοι οι πολίτες. Και επίσης ε, καταλογίζεται και ένα έγκλημα παρεμποδισμού στην πρόσβαση στις πληροφορίες. Επομένως, όχι μόνο δεν επέτρεψαν στους ανθρώπους να συμμετέχουν, αλλά και επίτηδες υπήρξε παρεμπόδιση ε, πληροφόρησης των πολιτών. Επομένως, ε, θέλω να σας ζητήσω να διατηρήσετε ανοιχτή αυτή την αναφορά και να πω στην Κομισιόν ε, ότι ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πως θεωρείτε ότι δεν υπάρχει παραβίαση της κοινωτικής νομοθεσίας εφόσον χρειάζεται εδώ μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για μια νέα για την έναρξη μια τέτοια δραστηριότητα. Υπάρχει εδώ ουσιαστική διαφοροποίηση ενό υφιστάμενου βιομηχανικού σχεδίου και αν δεν υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση για την επανέναρξη μιας ε, νέας εξορρεκτικής δραστηριότητας ε, καθώς ε, αυτές ε, αυτά τα λίμματα θα πάνε σε κάποιες ε, λίμνες και δεξαμενές που έχουν δημιουργηθεί το 39, τότε τι γίνεται εδώ. Έτσι λοιπόν γι' αυτό θέλω να διατηρηθεί η ανοιχτή αναφορά και πιστεύω ότι το αίτημα του αναφέροντα να υπάρξει αποστολή στην περιοχή είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σοϊντό. Ευχαριστώ. Καταρχήν, ε, να πω ότι άκουσα τον αναφέροντα. Είχαμε ε, μία σειρά χαρακτηρισμών που δεν ε, κατανοώ. Είχαμε απλώς ε, κάποιες δηλώσεις χωρίς καμία απόδειξη και εμένα μου δίνεται η απάντηση ότι δεν έχουμε ένα πολιτικό παιχνίδι πριν από τις επόμενες εκλογές. Εγώ είμαι υπέρ ότι πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά την εξορρυκτική δραστηριότητα. Όμως θα πρέπει να είμαστε αυστηροί, γιατί βρισκόμαστε εντός ενός νομικού πλαισίου και ουσιαστικού δικαίου, αλλά και σε ό,τι αφορά και τις διαδικασίες. Σας είμαστε αυστηροί, λοιπόν. Ας ε, σεβόμαστε την ε, διαδικασία, αλλά και τις ε, και τον νόμο, γιατί διαφορετικά νομίζω ότι θα ακολουθήσουμε λανθασμένη οδό. Και ακολουθώντα την ισχύουσα νομοθεσία, αυτό είναι ο δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε για να προσεγγίσουμε τα προβλήματα και να αφήσουμε τον πολιτικό πορτουνισμό. Με εξέπληξε ένα συνεγερμό ε, σήμερα το πρωί είναι σαν να ε, προσπαθούσαμε να καλύψουμε εδώ λίγο τα πράγματα. Κάποιοι μίλησαν ε, ότι μπορεί να υπάρχουν επιπτώσεις για την ε, καλλιέργεια των θαλασσινών. Κοιτάξτε, είναι ένα πολύ μεγάλο κλάδος, πολύ σημαντικός αυτός από κοινωνικό και οικονομικό, από οικονομική και κοινωνική σκοπιά. Θέλω να επικεντρωθώ στο θέμα γιατί προκύπτει ότι είναι ουσιαστικά ε, στα δικαστήρια αυτή η υπόθεση και επομένως ε, θα πρέπει να σεβαστεί η Επιτροπή Αναφορών ε, του χρόνου της δικαιοσύνης. Εδώ η κυβέρνηση της Γαλλικίας υπερασπίστηκε τη δράση της, αλλά υπερασπίστηκε και τον κατηγορούμενο. Όμως εμείς δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει μόνο ένα τεκμήριο δικαιοσύνης, ε, όχι μόνο στην Ισπανία, αλλά και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αρχές ε, της ε, Ανδαλουσίας σέβονται τις δικαστικές διαδικασίες και σήμερα συνεχίζει να είναι ανοιχτή η έρευνα. Γι' αυτό πιστεύω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να απόσχει από οποιαδήποτε δράση που θα μπορούσε να παρέμβει με την ποινική διαδικασία. Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι δεν ε, χρησιμοποίησαν ε, τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι αναφέροντες ε, στο εθνικό τους κράτος, ούτε ο αναφέρον, ούτε η Ένωση που προεδρεύει χρησιμοποίησαν την προσφυγή που προβλέπεται στον, στην περιβαλλοντική νομοθεσία κατά της επικαιροποίησης του σχεδίου που υιοθετήθηκε τότε. Γι' αυτό πιστεύω ότι η Επιτροπή Αναφορών δεν μπορεί να μετατραπεί στο δικαστήριο των 28 κρατών μελών. Εμείς δεν μπορούμε να φέρνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιες διαμάχες που θα πρέπει να επιλύονται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Και γι' αυτό επιμένω ότι η ύπαρξη της δικαστικής έρευνας ε, να αποτρέψει οποιαδήποτε αποστολή της ΠΕΤΗ στη Γαλλικία. Θα πρέπει να σεβαστούμε τους χρόνους της δικαιοσύνης και μία ερευνητική αποστολή θα μπορούσε να παρέμβει στη δικαστική διαδικασία. Και τέλος, ε, για την ουσία του ζητήματος. Ε, αφόσον εξετάζουμε τα έγγραφα, και εγώ χτες το βράδυ είδα το έγγραφο αυτό, Φαίνεται ότι δεν ε, είναι ακριβές να αναφέρουμε ότι ε, μιλάμε για νέο άνοιγμα του ορυχείου. Γι' αυτό το σχέδιο ε, ε, δεν θα χρειαζόταν απαραίτητα περιβαλλοντική αξιολόγηση αντικτύπου. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε για νέο άνοιγμα του ρηχείου γιατί τα δικαιώματα είναι από το 1800 ε, και το τελευταίο από το 1900. Έτσι λοιπόν ποτέ δεν έχει κλείσει ή εγκαταλειφθεί αυτό το ρηχείο. Και επομένω δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο της, ε, ε, του νέου ανοίγματο του ορυχείου. Σύμφωνα με την νομοθεσία υπήρξε μεταφορά του δικαιώματος που δεν αφορά την περίοδο ισχύως. Ε, η νομοθεσία που αναφέρει ο αναφέρον ε, δεν ε, μπορεί να εφαρμοστεί στο ρηχείο του Σανφίν. Και μιλώντας με πολιτικούς όρους, η δράση της σημερινής κυβέρνησης της Γαλλικίας υπό το Λαϊκό Κόμμα δεν διαφέρει καθόλου από τις δράσεις της τοπικής κυβέρνησης όταν κυβερνούσαν δύο κόμματα, γιατί από το 2008 ε, ε, ουσιαστικά τα δικαιώματα ε, για την εξορρυκτική δράση τα έδωσε η προηγούμενη κυβέρνηση που αποτελούνταν από δύο κόμματα. Γι' αυτό εγώ νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε τα έγγραφα της ε, αρμόδιας αρχής αλλά νομίζω ότι δεν είναι καθόλου σκόπιμο να έχουμε τώρα αποστολή στη Γαλλικία, κυρίως όταν υπάρχει εκκρεμής δικαστική διαδικασία. Και κανένας δεν πρέπει να παρέμβει. Και πόσο μάλλον μια πολιτική οργάνωση δεν πρέπει να παρέμβει στο έργο της δικαιοσύνης. Ευχαριστώ. κυρία Τόμ. Έχω τα εξή σχόλια στον τελευταίο ομιλητή. Δεν έχει υποχρέωση ο αναφέρον να προσφύγει σε τοπικό δικαστήριο. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να στείλει επιστολή σε μας. Ε, η πρότασή σας είναι πρόταση να καταργηθεί η Επιτροπή Αναφορών και να πρέπει οι άνθρωποι να αναφέρονται στο ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όχι, εμείς είμαστε σε άμεση επαφή με τους πολίτες και αυτός είναι ο ρόλος μας. Τώρα, η αναφορά υποβλήθηκε το 2017, όχι με την προηγούμενη κυβέρνηση. Για δύο χρόνια περιμένουμε απάντηση. Είμαι πρώην δημοσιογράφο. Η, αναφορά αυτή είναι πολύ καλογραμμένη, είναι πολύ σαφής και βασίζεται σε στοιχεία. Ωραία. Ο λόγος για δύο λεπτά στον αναφέροντα. Προ την Κομισιόν θα ήθελα να πω ότι εμείς οι καθημερινοί συνηθισμένοι πολίτε στη Γαλλικία δυσκολευόμαστε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου συστηματικές παραβιάσεις. Μοντενέμε, Σαντακόβα, Τόρο είναι άλλε περιπτώσει, Μας πήρε έξι χρόνια για να στήσουμε αυτή την ε, υπόθεση, να ε, ετοιμάσουμε τα στοιχεία μας. Πέρσι η γαλλικιανή κυβέρνηση ε, εξέδωσε μια οδηγία για την, τον περιοριστικό εφαρμο, ε, περιοριστική εφαρμογή της συμφωνίας του άρχους στην Ισπανία. Συστηματικά δυσκολευόμαστε να ε, αποκτήσουμε πρόσβαση σε οποιαδήποτε έγγραφα σχετικά με, την, με τα ορυχεία. Και πάλι παραβιάζεται η σύμβαση του άρχους. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Κύριε Σόιδο, σε ό,τι αφορά την έκθεση που, πήρατε χτες, που πήραμε χτες ε, και χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανένα, φανταστείτε αυτή η Επιτροπή να ζητούσε μια έκθεση για το Τσερνομπίλ για ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Και η κυβέρνηση έλεγε ότι δεν ε, παθεί τη ζημιά το Τσερνομπίλ, αλλά ένας αχυρώνας εκεί δίπλα. Αυτό συμβαίνει. Πρόκειται για φράγματα τα οποία χτίστηκαν ακριβώς για τη λειτουργία των ορυχείων. Τώρα κάποιοι προσπαθούν να το αρνηθούν και λένε ότι είναι υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Ε, δεν, δεν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα το πώς επηρεάζει τα, ε, της ρίας. Ε, έχουμε πριν από μερικά χρόνια μια έκθεση της με εμπειρογνώμονα και με συγκεκριμένα στοιχεία για σοβαρή μόλυνση από χαλκό, ε, ψευδάργυρο και κάδμιο στην εκβολή του Ρία, της ε, Ρίας Δεμόρος ε, στη Γαλλικία. Το 2018 υπάρχει ψήφισμα, ε, μάλλον απόφαση για την μεταφορά των δικαιωμάτων και σε αυτήν την απόφαση αναφέρεται ότι το σχέδιο θα πρέπει να ξανά κάνει η εταιρεία που τον αναλαμβάνει θα έπρεπε να ξανακάνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ποτέ δεν αμφισβητήθηκε αυτό, αλλά ξαφνικά η, ο όρο αυτό, η προπόθεση αυτή εξαφανίστηκε. Γι' αυτό λόγο γίνεται και ε, εισαγγελική έρευνα. Ζητούμε τη στήριξη του Κοινοβουλίου, τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να γίνει μια διαρευνητική επιτόπου επίσκεψη για να γίνει αντιληφτή η συστηματική παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας εκεί, η συστηματική παραβίαση των ευρωπαϊκών οδηγιών. Perfecto. Ωραία. Λέει η Πρόεδρος, ακούσαμε την Κομισιόν, ακούσαμε τις, ε, τις ε, ε, πολιτικές ομάδες των ετώντα. Θα αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή Χθε έφτασε η απάντηση της ε, Περιφερειακής Κυβέρνησης τη Γαλλικία, ε, χθε το βράδυ, ε, έφτασε και στην Κομισιόν. Η Κομισιόν δεν είχε χρόνο προφανώς να αξιολογήσει αυτές τις πληροφορίες, οπότε θα ζητήσουμε από την Κομισιόν μόλις το κάνει να μας υποβάλει μια έκθεση. Σε ό,τι διαφορά τις αποστολές, οι πολιτικές ομάδες γνωρίζουν πολύ καλά τη διαδικασία. Όποιος, όποιο, όποια πολιτική ομάδα θέλει μπορεί να ζητήσει να διενεργηθεί μια επιτόπια αποστολή. Αυτό προτείνω για, το, για τη συνέχεια που θα δώσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον αναφέροντα για την παρουσία του. Αυτό ήταν το τελευταίο μέρ, σε σημείο της ημερησίας διάταξης το πρωί. Οπότε θα κλείσουμε την συνεδρία αυτή και θα συνεχίσουμε στις 2.30. Αλλά βλέπω κυρία Άουκεν θέλει το λόγο κάτι πρόσθετο. Θα πρέπει να τοποθετηθούμε επί της θέσης της Κομισιόν ότι ε, ακόμα και αν υπάρχει παραβίαση του, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας δεν θα πρέπει να ασχολούμαστε με μονομένες περιπτώσεις. Δεν θα πρέπει να δεχτούμε αυτή την προσέγγιση. Πρόκειται για συστημικό πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά γενικότερα ε, είναι λάθος να πούμε ότι οι μεμονωμένες περιπτώσεις δεν αξίζουν την προσοχή μας. θα πρέπει να τηρήσουμε αυτό που κάνουμε παραδοσιακά και ιστορικά. Ακόμη και μονές περιπτώσει αξίζουν προσοχή. Πρόεδρος, κύριε Άουκεν, ο κύριος Σεύκοβιτς, αντιπρόεδρος και επίτροπος, ε, θα, ε, θα μας επισκεφθεί, ε, μας το υποσχέθηκε χτες και ήταν και δική του πρόταση μάλιστα, να έρχεται συχνά στην Επιτροπή Αναφορών Οπότε, μια και αναφέρεται κάτι πιο γενικό, καλύτερα να μας απαντήσει ο ίδιος ο Επίτροπος. Ωραία, κλείνουμε τη συνεδρία, θα τα ξαναπούμε στις 2.30.